προσεχώρησε, άψε το ΕΛΚ και προσεχώρησε στους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές. Η δεύτερη ανακοίνηση που θέλω να κάνω από το ECR έχω πάρει ανακοινώσεις για αλλαγές στον κατάλογο των αντιπροσωπιών. Ε, αυτός ο κατάλογος θα δημοσιευτεί και μέχρι τη δημοσίευση των πρακτικών ε, μπορείτε βέβαια να καταθέσετε ενστάσεις και όταν δημοσιευτούν πλέον δεν θα είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προχωράμε στην ψηφοφορία.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 Έχω ε, τη διαδικαστικό του κυρίου Νιούρεκ. Γιούρεκ, παρακαλώ κύριε Γιούρεκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρόεδρε, θα ήθελα βάσει του άρθρου 164 του κανονισμού να χρησιμοποιήσω τη δυνατότητα να απαντήσω σε κάποιες διαπιστώσεις, κάποια πράγματα που ακούστηκαν εναντίον μου. Ο κύριος Λάντορφ δεν δέχτηκε νωρίτερα να παρέμβω. Θέλω λοιπόν να απαντήσω στην κυρία Κουτρίσκα για αυτά που είπε κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρία Κουτρίτσκα. Η κυρία Κουτρίτσκα ε, ξεπλάγει για την αντίδρασή μου σε αυτά που άκουσα από το Συμβούλιο. Εγώ πιστεύω ότι το Συμβούλιο πρέπει να είναι πάντα εδώ κατά διάρκεια της συζήτησης για την μετανάστευση. Όσον αφορά το θέμα της εθελοντικής βάσης για την εφαρμογή των ποσοστώσεων, δεν ξέρω πού είναι ο πρόεδρος Τούσκ Ξέρω ότι ήταν στην προκλογική εκστρατεία στην Πολωνία αυτή τη βδομάδα, αλλά σήμερα έπρεπε να είναι εδώ, να βρίσκεται εδώ και στη συζήτηση αυτή να μιλάει εκ μέρους των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου, γιατί είναι η πρώτη του υποχρέωση αυτή και μετά έρχονται όλα τα άλλα. Η κυρία Κουτρίτσκα παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Επειδή ο κύριος Γιούρεκ αναφέρθηκε στο όνομά μου και στο πρόσωπό μου, θέλω και εγώ να απαντήσω σε αυτά που είπε. Το Συμβούλιο εκπροσωπήθηκε από την Υπουργό, την ασκούντα την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προετοιμάζει έτσι κι αλλιώς την εταιρική σχέση ε, που τη διάσκεψη αυτή δηλαδή που θα λάβει η χώρα αύριο και μεθαύριο στη Ρήγα. Οπότε τα σχόλια του κ. Γιούρεκ δεν